Πρόκειται για την προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για το θέμα των εξαγωγικών ελέγχων προϊόντων διτής χρήσης. Ο συντάκτης της ερώτησης, ο κύριος Μπέντ Λάγκη, έχει το λόγο πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν είμαι απλώς ο συντάκτης ως άτομο, απλώς είμαι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου και ως τι ούτως έχω θέσει αυτό το ερώτημα. Πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ένα είδος γραβιέρας, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προϊόντα δυτής χρήσεως. Είναι πολύ δύσκολο για μας να διαφοροποιήσουμε το κατά πόσο ένα προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει παραγωγή χάρη μια εργαλειομηχανή ή για να χρησιμοποιηθεί ως βάση εκτόξευσης ενός πυράβλου. Σε ό,τι αφορά το λογισμικό και τις τεχνολογίες επικοινωνίες, τα πράγματα είναι, πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. και είναι εκπληκτικό όταν κάποιοι ακτιβιστές στο Λονδίνο παίρνουν κάποιο mail στο οποίο έχουν ένα δούριο ύπο, έχουν δηλαδή ένα κακόβουλο λογισμικό το οποίο εξασφαλίζει ότι παρακολουθείτε το τηλέφωνό τους και όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν με το τηλέφωνό τους, το ευφυές τηλέφωνό τους να μπορούν να την χάνουν ανάγνωση από τρίτους. Και το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς χώρους για να υπάρξει όχι επικοινωνία, αλλά παρακολούθηση ακτιβιστών, πολιτικών αντιπάλων, ατόμων που είναι αντιφρονούντες και των οποίων παραβιάζονται με αυτόν τον τρόπο τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι λοιπόν απαραίτητο ότι δεν πρόκειται μονάχα για τους ε, ακτιβιστές κρατών που ζουν σε καθεστώτα τα οποία δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ενδεχομένως και τρομοκρατικά καθεστώτα να μην παίρνουν αυτές οι χώρες τέτοια <clears throat> προϊόντα διτής χρήσης, αλλά επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το λογισμικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται και στην Ευρώπη από τρίτες χώρες για να παρακολουθεί τους πολίτες και τους ε, ακτιβιστές. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα σε χώρες όπως είναι το Μπαχρέιν, όπως είναι το Ιράν, όπου δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό σύστημα με ευρωπαϊκή τεχνολογία ή στη Συρία ή στην Λιβύη όπου οι μυστικές υπηρεσίε αγόρασαν μια επιχείρηση της οποίας το σύνθημα είναι με τον καλύτερο και τον απλούστερο τρόπο παρακολουθούμε. Και φαίνεται ότι αυτή η εταιρεία έχει 50% μερίδιο αγοράς στην Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι η Αιθιοπία, η Νιγερία, το Κατάρ είναι χώρες οι οποίες δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ακολουθούν κατά γράμμα τις ευρωπαϊκές ε, αρχές και αξίες, αυτές οι χώρες παίρνουν τέτοια προϊόντα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να σκεφτούμε και ότι με την ε, Συμφωνία της Βασιλείας το 2013 το λογισμικό ιδούρι ύπη και ελεκτικού χαρακτήρα λογισμικό ε, στα αγαθά αυτά που πρέπει να είναι στοιχεία υποκείμενα σε ελέγχου διτής χρήσης. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία, καμία διάταξη που εξασφαλίζει ότι το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακόβουλους σκοπούς και να χρησιμοποιηθεί από αυτούς οι οποίοι θέλουν να παρακολουθούν και να σπιουνάρουν τον πληθυσμό τους. Και φυσικά όλα αυτά έχουν διαστάσεις στρατηγικού χαρακτήρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τρία ερωτήματα προς την ε, κυρία Πίτροπο. Τι γίνεται καταρχήν με την ενι, ενιαία και αποτελεσματικό, την ενότητα και την αποτελεσματικότητα των εγκρίσεων αγαθών διτής χρήσης. Τι κάνουμε ή εγκρίνονται τα πάντα. Πώς δρούμε για να μην τα δίνουμε αυτά σε περιοχές εμπόλεμες. Δεύτερον, το θέμα του ελέγχου. Ο έλεγχο λέτε ότι είναι μονάχα εξ και όχι εκ των προτέρων. Μόνο εκ των υστέρων ξέρουμε ποια αγαθά έχουν εξαχθεί σε, πώς, ε, σε ποια χώρα. Και τότε είναι πολύ εύκολο να υπάρξει κατάχρηση αυτών των ε, εξαγωγών. Και φυσικά Εκεί λαμβάνει υπόψη και τα εμπορικά συμφέροντα. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απάντησή σας σε όλα αυτά. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει η Επιτροπή Μάλμστρομ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητοί βουλευτέ, και χαίρομαι που έθεσατε αυτό το πολύ σημαντικό αλλά και δύσκολο θέμα. Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικό παραγωγό ε, τέτοιων και εξαγωγέα ε, ε, προϊόντων διπλή χρήση. Η εξ, έλεγχη, εξαγωγική έλεγχη είναι βασικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τι εξαγωγές, 14 δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά του ελέγχου. Είναι σημαντικό και για την διεθνή ασφάλεια. Το καθεστώς ε, για τους ελέγχου έχει σταδιακά αυξηθεί τα τελευταία δεκαετία. Περιλαμβάνει ένα στεναρό πλαίσιο, μοντέλο για τρίτες χώρες, αλλά φυσικά ο κόσμος μεταβάλλεται και δεν μπορεί να παραμείνει στατικό το μοντέλο αυτό. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί, να αναθεωρηθεί για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσει που έχουν μεταβληθεί. όπω ανέφερε και ο κ. Λάγκε, θα πρέπει να υπάρχουν σύγχρονε λοιπόν ικανότητες ελέγχου σε ό,τι αφορά το κοινωτικό εμπόριο και πέρα του κοινωτικού εμπορίου. Σύμφωνο με τι ανησυχίε που εκφράστηκαν σε ό,τι αφορά την ε, τεχνολογία παρακολούθηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε, έχουμε προτείνει νομοθεσία προ την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε εγκρίνει τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους ε, πράξη κατά εξουσιοδότηση για να εφαρμοστούν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο οι πολυμερείς ε, διατάξεις της Συμφωνίας του Βασανάρ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Επίσης, η εξαγωγή τεχνολογίας παρακολούθηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, αναθεώρησης της πολιτικής εξαγωγών. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του περσινού έτους δημοσίευσε ανακοίνωση όπου αναφέρει τέτοιους ελέγχους και θα αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε κάθε περίπτωση τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξαγωγίες. Να δημιουργηθεί, για παράδειγμα, ως όρος τα ανθρώπινα δικαιώματα για περαιτέρω ελέγχους και για άρνηση εξαγωγών. Αλλά φυσικά θα πρέπει να ζυγοσταθμίσουμε τις απαντήσεις μας και την ανταπόκριση μας. Θα πρέπει να δούμε ποια αντικείμενα, ποια προϊόντα αποτελούν ε, επικίνδυνα προϊόντα και να έχουμε υπόψη ότι κάποια από τα προϊόντα αυτά έχουν και νόμιμες χρήσεις. Να μην ξεχάσουμε ότι ενδεχομένως και προϊόντα από τρίτες χώρες να έρθουν να αντικαταστήσουν τα δικά μας προϊόντα. Αυτό θα βλάψει και την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και την, ε, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσπαθούμε να προωθήσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να προσαρμόσουμε τον κανονισμό Θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε συμπράξεις μεταξύ των διαφόρων ελέγχων ασφαλείας. Και αυτό είναι μόνο ένα μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, για παράδειγμα, να στοχεύσουμε συγκεκριμένες χώρες. Και αυτό καλύπτεται από το άρθρο 250 της συνθήκης, ό,τι φάση της κυρώσης. Όπως ξέρετε, η ανακοίνωση δίνει και ένα όραμα για το μοντέλο για να υπάρξει ανάπτυξη των σχετικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, προκειμένου να είναι μεγαλύτερη η αποδοτικότητα των ελέγχων και να ελαχιστοποιηθεί η στρέβλωση της αγοράς, προκειμένου να υπάρχουν ίσοι όροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις τρίτες χώρες. Για παράδειγμα, ανεκτή αδειοδότηση, για να μην υπάρχει καθυστέρηση των εξαγωγών και έλεγχη εξάντα για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα. Αυτό θα περιορίσει και το κόστος αλλά και τις καθυστερήσεις των ελέγχων και παράλληλα θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλεια. Συμφωνώ με το Κοινοβούλιο ότι η τεχνική φύση των προϊόντων αυτών σημαίνει ότι θα πρέπει να, συμμετέχει, να συμμετέχουν ε, εμπειρογνώμονες. Γι' αυτό λοιπόν ε, κινητοποιούμε εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν ε, αναθεώρηση των ελέγχων μας προκειμένου να είναι σίγουρο ότι είναι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα ήθελα να τονίσω ότι ο εθνικός κλάδος είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πραγματικά συμπράξη μαζί του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Και τώρα από τι πολιτικέ ομάδε, πρώτον Πρώτος από το έλεγχο, ο κύριος Σάινφελτ. Δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο έλεγχος του διεθνούς εμπορίου συγκεκριμένου τύπου προϊόντων, προϊόντων τα οποία μπορεί να έχουν διπλή χρήση, είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολα παρά επανειλημμένους έλεγχους να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην χρήση των προϊόντων. Η τεχνολογία είναι πλέον κάτι το καθολικό και εξαρτάται τελικά από την χρήση την οποία θα κάνει ο τελικός χρήστης. Ένα άλλο θέμα είναι και το θέμα της μετοχής των μικρομεσαίων το διεθνές εμπόριο. Αυτό είναι κάτι το θετικό. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι η βάση του οικονομικού συστήματος και δεν θα πρέπει να τις επιβαρύνουμε με την γραφειοκρατία και επιπλέον κόστη. Πρέπει ε, να δούμε τις ανάγκες που έχει το διεθνές εμπόριο και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να βρούμε ένα σωστό σύστημα ελέγχου της εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται για την παράνομη καταστολή των εκδηλώσεων των πολιτών σε διάφορες χώρες και περιοχές. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε το θέμα της ανάπτυξης της έρευνας. Πάντως δεν θα πρέπει να θίξουμε σε καμία περίπτωση την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρεμποδίσουμε την έξοδο των μικρομεσαίων στις διεθνείς αγορές. Ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος Λάιχτ Φρίδ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Μερικές φορές είναι κουραστική η πολιτική. Πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει τις λεπτομέρειες και αυτό κάνει ακόμα πιο εργόδια όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι ο πρώτος βέβαια ο οποίος έχει αντιμετωπίσει το θέμα των αγαθών διπλής χρήσης. Αλλά πρέπει να εξηγήσω ίσως τι ακριβώς γίνεται με τα αγαθά αυτά που δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης, ίσως και την κοινή γνώμη. Δίνουν τη δυνατότητα όμως τα αγαθά αυτά ορισμένοι να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη με μεγάλη ευκολία. Λοιπόν, ουσιαστικά πρόκειται για όπλα, πρόκειται για επικίνδυνα όπλα. Θυμάμαι τον Επίτροπο Ντεχούχτ, ο οποίος είχε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά εσείς κύριε Επίτροπε πιστεύω ότι θα μπορέσετε να δώσετε την απαραίτητη σημασία στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τομέα αυτό. Καταρχήν υπάρχει η έλλειψη, <clears throat> η έλλειψη ισότητας ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Βλέπω τον κύριο Ντάρτμουθ, ο οποίο είναι κρυμμένος πίσω από τη σημεούλα του. Έχουμε έθνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες εξαγωγών, ενώ κάποια άλλα δεν έχουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ αυστηρούς κανόνες και νοιάζεται για αυτούς τους κανόνες. Υπάρχουν άλλε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν τέτοιου κανόνε. Και επομένω βρίσκεται σε μειονεκτική θέση το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτήν την περίπτωση. Πιστεύω ότι ο κύριο Δάρκου θα συμφωνούσε με, μαζί μου. Αυτή είναι μια κατάσταση που χρειάζεται να αλλάξει. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκού κανόνε οι οποίοι να είναι κοινοί. <clears throat> Δεύτερον, θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα. Τι καλύπτεται από, τα, από τους κανόνες αυτούς υπάρχει ένας κατάλογος και ότι δεν είναι σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να εξαχθεί. Αλλά είναι αυτή η σωστή αντιμετώπιση. Και ένα δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε είναι το θέμα των εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων <clears throat> ελέγχων. Η εκ των προτέρων ε, εξέταση κοστίζει περισσότερο σε χρήματα. Η εκ των υστέρων όμως κοστίζει πολύ περισσότερο σε ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μοναχα το κόστος των επιχειρήσεων. Και υπάρχει όπως αναφέρθηκε το θέμα του software που πολλά από αυτά τα αγαθά είναι αγαθά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις ε, Ηνωμένες, στο, στη Μέση Ανατολή έχουν ε, εξαχθεί πάρα πολλά στοιχεία software τα οποία έχουν οδηγήσει στην απώλεια πάρα πολλών ζώων. Σας ευχαριστώ κύριε Λάιφτιτ για τον ε, Earl of Dartmouth έχετε χρόνο ομιλίας. Ε. Γι' αυτό λοιπόν ε, αυτά που θέλετε να κάνετε με την μπλε κάρτα καλύτερα να τα κάνετε στην χρονομιλία σας. Ευχαριστώ. Φωτίγκα από το ECR. I was Αναφέρθηκα ιδιαίτερω από τον ομιλητή με πολύ φιλικό τρόπο και ήθιστε να μπορώ να απαντήσω 30 δευτερόλεπτα. Επίσης ήθιστε, λέει ο πρόεδρος, ο πρόεδρος να λαμβάνει την απάντηση, να λάβει την απόφαση αυτή. Και ήθιστε, αν ο μιλητής που ζητά μπλε κάρτα έχει χρόνο ομιλίας, να μην έχει, να μην παίρνει το λόγο. Η συνάδελφος Άννα Φωτίγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, κάποιες χώρες όπως είπα, ο Καναδάς το Μαρόκο έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και έχουν συμπεριλάβει τον χώρο της τεχνολογίας στις κυρώσεις αυτές. Εμείς αποφασίσαμε διαφορετικά. Οι δικές μας κυρώσεις δεν καλύπτουν το ευρωπαϊκό, πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα. Οι εμπορικοί λοιπόν δορυφόροι της ε, Airbus και του Galileo ε, εκινήθηκαν τρεις φορές και χρησιμοποιήθηκαν το Σόγιος και το Πρωτέους. Με καταστροφικά αποτελέσματα. Τα βλήματα οι δορυφόροι μάλλον, δεν ε, πήραν σωστή τροχιά. Ποιος ε, φταίει λοιπόν για, τα, για τις αδυναμίες, τα προϊόντα της ε, χρήσης ή η έλλειψη αλληλεγγύης από πλευρά των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ε, επίθεση στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Η Ρίτσια Σχάκε από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, Επίτροπε. Σήμερα μας υπενθυμίζουν ε, το τι διακυβεύεται στη συζήτηση αυτή. Οι hacker, ε, οι οποίοι ε, έχουν σκοπό να κλέψουν, να υποκλέψουν ε, δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε, τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από software. Οι εξαγωγές ε, συμπεριλαμβάνονται στο Toxnet, όπου έγινε επίθεση πριν από κάποια χρόνια και όπου βρέθηκαν χώρες όπως το Ιράν, το Μεξικό και Συχνά αναζητώμε τους υπέτειους στην Κίνα και στη Ρωσία, αλλά τα συστήματα αυτά μπορεί να έχουν κατασκευαστεί και στην Ευρώπη. Ακόμα και αν έχουν αναπτυχθεί για τις μυστικές υπηρεσίες, οι τεχνολογίες αυτές ε, διαδεύονται πάρα πολύ, γίνονται όλο και πιο φθηνές, όλο και πιο εύκολες στη διάδοση. Φανταστείτε λοιπόν τους ε, μη κρατικούς φορείς να δρουν στον κλάδο αυτό για την παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παραβίαση των υποδομών μας και των ευάστητων δεδομένων. Αυτά τα δισεκατομμύρια ψηφιακών όπλων μπορεί να αποτελέσουν το μεγαλύτερο μπούμερανγκ που έχουμε δει ποτέ. Και θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε τα κενά στην νομοθεσία μας και τα συστήματα μαστικής παρακολούθησης και υποκλοπής χωρίς νομική βάση και χωρίς συνένεση θα πρέπει να εξετάσονται πολύ πιο στενά. Χρειαζόμαστε διαφάνεια. Ε, υπευθυνότητα όρους έγκρισης και αδειοδότησης και ίσους όρους για όλους τους φορείς και όλες τις επιχειρήσεις. Επίτροπε, θα παρουσιάσετε θετικό ή αρνητικό κατάλογο χωρών για τις τεχνολογίες αυτές και πώς θα ανταποκριθείτε στις κρίσεις. στην κρίση αυτή θα υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός. Καλή ιδέα θα ήταν. Επίσης, ε, να γίνει μέτρα εκτύπου στη φάση έρευνας και ανάπτυξης για να ξέρουμε τι μπορεί να κάνουν τα προϊόντα αυτά θέλουμε ευφυή νομοθεσία, το συντομότερο δυνατόν και πολύ περισσότερα από αυτά που ενέκρανε το Συμβούλιο την Παρασκευή, γιατί αν περιμένουμε κι άλλο η κατάσταση θα μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους, πρασίν, για τους ε, αριστερούς η κυρία Μινέωρ για 1,5 λεπτό. Αλλά δεν είναι παρούσα. Πάμε στους πράσινους και δίνουμε το λόγο στην κυρία Σκα Κέλλερ για ένα λεπτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει τα αγαθά τα οποία μπορεί να φαίνονται ότι είναι άκακα αλλά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραδείγματος χάρη για την παρακολούθηση ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι να προστατεύσουμε τους, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Αυτό λοιπόν δεν <clears throat> είναι αρκετό να ελέγχουμε εκ των υστέρων τα, τα αγαθά έχουν φτάσει ήδη στα λάθο χέρια. Χρειαζόμαστε ελέγχου εξάντε και όχι εξ Και όσο εξελίσσεται η τεχνολογία όλο και περισσότερο πρέπει και εμεί να εξελίξουμε τη δική μα νομοθεσία. Υπάρχουν οι τεχνολογίες παρακολούθησης οι οποίες μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό και δεν μπορούμε να τις εξαιρούμε από αυτή τη διαδικασία. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει τώρα να κάνει κάτι για όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε ήδη το 2015 μια πρόταση. Δεν πρόκειται για ένα καθαρά τεχνικό θέμα είναι θέμα προστασίας των ανθρώπων και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Αμεσής Δημοκρατίας ο κύριος Βίλιαμ Ντάρτμουθ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παδέ εν ώψη του ότι έλαβε χώρα αυτή η ανταλλαγή. Διερωτώ με γιατί οι πολιτικοί που θεωρούν αυτούς φιλελεύθερους να είναι στην ουσία τόσο κατά της ελευθερίας. Ο κύριος Φερχόφστατ σαν παράδειγμα, ακούσαμε αυτά που έλεγε νωρίτερα και στην ουσία μιλάει με έναν τρόπο ο οποίος είναι καταχρηστικός και υβριστικός και όχι ε, δεν μεταφέρει επιχειρήματα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η συνάδελφος εκ δεξιών δεν είναι μέλος της ε, πολιτικής μου ομάδας, όπως πιστεύετε κύριε Πρόεδρε, να σας ενημερώνω καλύτερα την άλλη φορά. Η κυρία Φώτιγκα δεν ανήκει. Το Ηνωμένο Βασίλειο, εν πάση περιπτώσει, εφαρμόζει τις δικές του απόψεις στα θέματα καθορισμού του τι εξάγουμε και τι δεν πρέπει να εξάγουμε και γενικά σεβόμεθα το δικαίωμα των άλλων χωρών να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της δικής τους κυβέρνησης για τα εξαγώγημα ή μη προϊόντα και αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποφασίζεται από τους μη άμεσα εκλεγμένους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. οι επιχειρήσεις και οι εξαγωγείς για όλα τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αντικειμένων ειδών ε, διπλής χρήσης πρέπει να ζητούν την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι παράλογο. Το πλαίσιο της διπλής χρήσης στην ουσία δίδει περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως είναι ηγέτης εμπορικά δύναμη στον κόσμο για εκατοντάδες χρόνια και το καθεστώς αυτό της διπλής χρήσης της Επιτροπής είναι απαράδεκτο. Ζητώ συγνώμη στην κυρία Φώτιγκα θεωρώντας ότι ανήκει στην πολιτική σας ομάδα. μου, επόμενος ομιλητής. Επίτροπε, η εξαγωγή τεχνολογιών και προϊόντων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για, με διπλό τρόπο είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, τα αντικείμενα αυτά, τα ίδια αυτά πολλές φορές χρησιμοποιούνται εναντίον της ελεύθερης έκφρασης. Θα πρέπει λοιπόν οι μηχανισμοί εξαγωγών να είναι ε, σύγχρονοι και αποτελεσματικοί. Αυτό πρέπει να καλύπτει και τον δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό άπτεται και του θέματος της μεταφοράς των τεχνολογιών γενικότερα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον προηγούμενο Απρίλιο νομίζω υπογραμμίζει τις ελλείψεις και χαράζει ένα σωστό δρόμο για το μέλλον. Το θέμα είναι λοιπόν να στηρίξουμε και να επιταχύνουμε την εφαρμογή της πρότασης που τίνει στην ενίσχυση των ρυθμίσεων για τα προϊόντα διπλής χρήσης. Παράλληλα, ε, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πάρουν τα απαιτούμενα μέτρα. Δυστυχώς η σωστή χρήση ή η καταχρηστική χρήση αυτών των προϊόντων είναι ένα θέμα το οποίο κυρίως θα ελέγχεται από τα κράτη-μέλη. Αν τα προϊόντα αυτά πέσουν στα χέρια καταπιεστικών καθεστώτων είναι κάτι το οποίο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε να γίνει κάτι τέτοιο για λόγους κινησμού ή πραγματισμού έτσι ώστε μόνο να εξάγονται τα προϊόντα μας. Και εδώ και το θέμα των κυρώσεων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρες όπως η Ρωσία. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε η ασφάλεια, όπως λέγεται να μην επηρεαστεί από την κακή χρήση της. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ να μην ξεπερνάτε το χρονομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μόσκα. Πρόεδρε, κυρία Μάλστρομ, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προϊόντων διπλής χρήσης. και ε, λόγω της τάσης που υπάρχει για εντατικοποίηση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και λόγω της αυξημένης δυνατότητας και επιχειρησιακής ικανότητας των ε, τρομοκρατικών ομάδων. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δώσουμε τη μέγιστη δυνατή πρόσοχη στην ρύθμιση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προϊόντα διπλής χρήσης και θα πρέπει να επιταχυνθεί η αποδοχή της νομοθετικής πρότασης. Υπάρχουν όμως κάποιες ανησυχίες οι οποίες θα πρέπει να τεθούν. Θα πρέπει καταρχάς να λάβουμε υπόψη ε, την δυνατότητα ε, περιορισμού των απειλών της χρήσης των προϊόντων αυτών με μη σωστό τρόπο. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να δημιουργήσει ε, μια στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος ανώλων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν σε χώρες οι οποίες ε, δεν είναι τόσο διαφανείς. Η έλεγχοι θα πρέπει να είναι αυστηροί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και θα πρέπει ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στο ευρωπαϊκό εμπόριο, βλέποντας ποια είναι τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για τους ευαίσθητους τομείς. Και τελευταία ερώτηση είναι πώς μπορεί να υπάρξει μια κοινή ρύθμιση και κοινά στάνταρτς για την εξαγωγή των προϊόντων αυτών. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και εσάς αγαπητοί Δερμηνείς ευχαριστώ. Επομένως, ο μιλητής ο κ. Πρέτσελ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλάμε για τη τεχνολογία παρακολουθήσεις και η διπλή χρήση σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα σαφή στόχο, έχει ένα σαφή στόχο. ένας είναι ο στόχο, ένα είναι ο σκοπό χρήση. Κάθε φορά που συναντιόμαστε εδώ στο Στρασβούργο, το Κοινοβούλιο τη Πέμπτη ασχολείται με παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Και στι πιο πολλέ περιπτώσει διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιούνται τεχνολογίε παρακολούθηση, οι οποίε σε κάποιε περιπτώσει προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι περιπτώσει λοιπόν αυτέ, όπου πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα χρειαζόμαστε ε, έλεγχο εξάντε. Χρειαζόμαστε ένα κατάλογο για τις χώρες αυτές. Και θέσατε κάποια ερωτήματα. Είπατε ότι και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θύματα τέτοιων μυστικών υπηρεσιών. Τι περιμένετε από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν εξαγάγει μόνο προϊόντα, αλλά και τα δεδομένα των προϊόντων της. Τραπεζικά δεδομένα, ταξιδιωτικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ, Διακόπτη Πρόεδρος. Ο κύριος Τσεβάιος είναι ο επόμενος. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω απαντήσει σε κάποια από τα ερωτήματα που ήθελα να ρωτήσω στην Κομισιόν. Θα ήθελα να εστιάσω λοιπόν σε αυτό το οποίο ε, έχει γίνει για την βελτίωση και την ε, αναβάθμιση των κανόνων. Λέτε ότι θα συμπεριληφθεί στο μέλλον ο εξοπλισμός για την παρακολούθηση τελεπικοινωνιών. Αλλά αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό για ορισμένε χώρε. Και το ίδιο για ορισμένε υπηρεσίε συμβούλων. Πρέπει να έχουμε μια ε, ρύθμιση η οποία δεν κοιτάζει μοναχά το προϊόν αλλά και τη χώρα που είναι ο αποδέκτης αυτού του ο εισαγωγέας. Είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε ένοπλες διαδικασίες, είναι δημοκρατική χώρα ή όχι. Αυτά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα σε ένα ρευστό κόσμο. Θα πρέπει να μάθουμε λοιπόν από τα λάθη που έχουν κάνει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πουλήσαν αυτόν τον εξοπλισμό σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρήσει τι βασικέ αξίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας ακόμα και αν αυτό δεν βοηθάει τη βιομηχανία της. Πρέπει να προστατήσουμε πρώτα τα ανθρώπινα όντα. Ελπίζω λοιπόν ότι η πρόταση Κομισιόν θα πάει προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιγκίν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα προϊόντα αυτά είναι για πολιτική χρήση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικά όπως στα ανταλλακτικά της αεροναυπηγικής. Είναι η λεγόμενη διπλή χρήση. Εδώ μιλάμε για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς. Με συγχωρείτε πρέπει να σας διακόψω. Πρέπει να μιλάτε πιο αργά. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να γίνει διερμηνία λάβετε υπόψη και τους διερμηνείς. Ξαναρχίζω λοιπόν. Έλεγα ότι δεν μιλάμε για όπλα, αλλά για μέσα, για πολιτικούς σκοπούς. Άρα δεν υπάρχουν οι ίδιοι περιορισμοί, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει παραβίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό μιλάμε για την ε, τον, την ανθρώπινη, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις συμβάσεις που έχει προσπογράψει η Ευρώπη, απ' την άλλη όμως αναπτύσσει όπλα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι το 2013 στην ουσία πουλήσαμε χημικές ουσίες στη Συρία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Άρα Χρειάζεται καλύτερος έλεγχος των κρατών μελών, ιδιαίτερα για τα προϊόντα διπλής ε, χρήσης, έτσι ώστε να ξέρουμε τι χρήση πραγματικά γίνεται. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη έτσι ώστε η τεχνολογία Made in Europe να ελέγχεται όπως έγινε κατά τη διάρκεια της ε, Αραβικής Άνοιξης. Γι' αυτό θα ήθελα η Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες για τα προϊόντα διπλής χρήσης για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση όπως είπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τεχνολογικά προϊόντα και θα ήθελα να ελέγξουμε την εφαρμογή του κανονισμού από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα για αυτά τα προϊόντα διπλής χρήσης. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ενάμιση λεπτό, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ, η χρήση των προϊόντων αυτών μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδότηση παραγωγής όπλων, κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλο και περισσότερα συμβάντα καταπίεσης ε, χρησιμοποίησαν ε, τεχνολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ελέγχονται. Έτσι τώρα θα πρέπει να κλείσουμε κενά στο, στη λειτουργία του εμπορίου. Θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία και να εφαρμόζεται καλύτερα. Για να χρησιμοποιούνται σωστά αυτά τα προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ελέγχει τις εξαγωγές, τη διέλευση, ε, τη χρήση αυτών των προϊόντων ε, ως πολιτική κλειδί για την ασφάλεια, για την ειρήνη. Είναι στο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε την τεχνολογία και το λογισμικό της Ένωσης, ούτω ώστε να μην ε, εκτρέπεται από την θεμητή χρήση τους και η ψηφιακή υποδομή της Ένωσης όπως και τα συμφέροντά της σε στρατηγικό επίπεδο να διαφυλάσσονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός παίκτη σε αυτό το τομέα διεθνώς. Ω θεματοφύλακα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της ε, πολιτικής και της νομοθεσίας να υπάρχει παρακολούθηση του εμπορίου στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, διεθνείς προσπάθειες ελέγχου του εμπορίου σε αυτά τα προϊόντα είναι ξεπερασμένα και πρέπει να αναπροσαρμοστούν στο σύγχρονο κόσμο. Εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε. Είχα την εντύπωση ότι είχα δύο λεπτά, ενάμιση λεπτό λέει εδώ. Ευχαριστώ πολύ, σαφώς είσαστε. Ε, ευχαριστώ ε, ο κύριος Φερνάντες για λεπτό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρόθεση της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως δεν βρούμε επιμελώς έναντι των καταχρήσεων των κυβερνήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογικά προϊόντα ή λογισμικό δήθεν για πολιτικούς σκοπούς που δυστυχώς διονύζουν τα όπλα μαζικής καταστροφής. Λάβαμε υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική με βάση τα χάσματα που υπάρχουν. Έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει σοβαρές συνέπειες και μπορεί να έχει ακόμα περισσότερες. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τεχνολογίες και λογισμικό που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιούνται από τις αστυνομικές αρχές ή στρατιωτικές αρχές για την καταστολή ή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε μία ε, Ευρωπαϊκή Ένωση σύγχρονη αλλά και ευέλικτη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το τελικό μας χρονοδιάγραμμα με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής τον Απρίλιο. Χρειαζόμαστε όμως έναν, μια σαφή δέσμευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Νίκολα Ντάντι για ένα λεπτό. Grazie Presidente, signor Ευχαριστώ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα προϊόντα διπλής χρήσης δεν θα πρέπει να διέπονται από τους ίδιους κανόνες όπως ισχύει για άλλους παραγωγικούς τομείς. Χρειάζεται ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να υποπτεύσει τους πολίτες και τις κυβερνήσεις. Ιδιαίτερα σε έναν κόσμο που μεταλλάσσεται όλο ένα και περισσότερο και μετασχηματίζεται και μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας των λαών. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου και θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση αντικτύπου, μια προγενέστερη ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια αυτής της παραγωγής. Ελπίζω η Επιτροπή να φτάσει σε μία σύγκληση του, του ρυθμιστικού πλαισίου. Ένα λεπτό από εδώ και πέρα για όλους. Νικόλ Καπούτο. Να προλάβουν όλοι να μιλήσουν. Νικόλα. Ευχαριστώ. Χρειάζονται πιο σοβαροί έλεγχοι στην εξαγωγή αυτών των προϊόντων διπλής ε, χρήσης και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφαλή διαβίωση των πολιτών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εξαγωγές ε, τεχνολογίας διπλής ε, χρήσης προϊόντων που παράγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διτό σκοπό και, για, και οδηγούν και στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει ε, τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν, αλλά να υπάρχει ένα σύστημα κοινοποίησης εξάγκτε για αυτά τα προϊόντα διπλής χρήσης και θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια έτσι ώστε να πληρώσουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ και συνάδελφε. Ιβάν Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Το δίλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι δύσκολο να λυθεί. Είμαστε υπέρ περισσότερων κερδών που είναι θεμητό ή πράγματι υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα υπόλοιπα που παραβιάζονται τόσο συχνά σε χώρες εταίρους μας και που χρησιμοποιούν προϊόντα διτής χρήσης. Ακόμα παραπάνω τέτοια προϊόντα συχνά χρησιμοποιούνται εναντίον μας, εναντίον των πολιτών μας ή κατά των γειτόνων και φίλων μας Επομένως, φυσικά εγώ είμαι υπέρ της ιδέας να σκεφτούμε πρώτα τις ευρωπαϊκές αξίες τι οδήγησε στη δημιουργία του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μαριάς. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε η έλεγχη στις εξαγωγές προϊόντων διπλής χρήσης αποτελεί μια σημαντική δράση που πρέπει να ενθαρρύνει η ευρωπαϊκή ένωση και αυτό μπορεί να γίνει και στο διεθνές πεδίο με μηχανισμούς υιοθέτησης κοινών πρακτικών γνωστών και ως καθεστώτα ελέγχου εξαγωγών. το θέμα της προσχώρησης νέων μελών στα καθεστώτα ελέγχου εξαγωγών πρέπει να εξετάζεται με τεχνικά κριτήρια και να μην αποτελεί πεδίο άσκησης πολιτικών αποκλεισμού στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η τουρκία εμποδίζει την υποψηφιότητα της κύπρου στο καθεστώς ελέγχου πυραυλικής τεχνολογίας mtsr στον διακανονισμό βασεναρ και στην επιτροπή zanger. για το λόγο αυτό η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να στηρίξει την κυπριακή υποψηφιότητα στα εν λόγω καθεστώτα ελέγχου εξαγωγών ασκώντας πιέσεις στην τουρκία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ο συνάδελφος Ζωάν Φεραέρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Επίτροπε, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε εδώ τους ε, ελέγχους της εξαγωγές ειδών διπλής ε, χρήσης. Μιλάμε για τεχνολογίες και λογισμικό που χρησιμοποιούμε στις επικοινωνίε αλλά υπάρχουν και άλλες χρήσεις αυτής της ε, τεχνολογίας δήθεν για πολιτικούς σκοπούς. Στην ουσία γίνεται στρατιωτική χρήση. Γι' αυτό χρειάζεται μια νέα προσέγγιση, μια πιο διευρυμένη προσέγγιση. Μιλάμε για τα σχέδια, τα ερευνητικά σχέδια που διεξάγονται μαζί με τις αεροδορυφαρικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι σφαγές της Γάζας δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν χρησιμοποίησαν αυτή την τεχνολογία. Γι' αυτό θα πρέπει να μην έχουν πρόσβαση ορισμένες χώρες στη χρηματοδότηση τέτοιων ε, σχημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος Μάλμστρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για τη συμβολή σας στην πολύ ενδιαφέρουσα και σύνθετη συζήτηση Όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολλά τα προϊόντα που μπορούν να, χρησιμοποιούν για, να χρησιμοποιούνται για καλό σκοπό, αλλά συνεπάγονται και κινδύνους. Ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν καμιά φορά για παρακολούθηση ή για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να το δούμε αυτό. Ο έλεγχος των εξαγωγών δεν είναι ο μόνος τρόπος, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Προσπάθησα να πω ότι κάναμε κάποια πράγματα και τώρα ακούμε πολύ προσεκτικά τους πάντες για να αναβαθμίσουμε και να αναθεωρήσουμε την ε, νομοθεσία μας. Υπάρχει ανακοίνωση, υπάρχουν κάποιες ιδέες εκεί, ακούμε πολύ και τη βιομηχανία, τα κράτη-μέλη, αυτά που λέτε εσείς και βέβαια διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις πολύ δραστήριες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι δεν υπήρχε θέμα εδώ πριν από λίγα χρόνια. Τώρα υπάρχει, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουν τροποποιηθεί οι κανονισμοί, οι, πολιτικές βελτιώθηκαν, είναι ενήμεροι, ενήμερος ο κόσμος, αλλά χρειάζονται κι άλλα. Είναι σύνθετο το θέμα. Πρέπει να προχωρήσουμε σωστά, ούτω ώστε ο στόχος μας να πραγματοποιηθεί. Να, παράλληλα να μην ζημιώσουν οι εξαγωγές μας. Ε, όταν πάνε για καλό σκοπό. Τώρα λοιπόν ξανά είδαμε την νομοθεσία, είδαμε πολλούς, ακούσαμε εμπειρογνώμονες, εμπλεκομένους και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια προσεκτικά ισορροπημένη πρόταση που θα την υποβάλλουμε του χρόνου και προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε αυτή την προσπάθεια και θα χαρούμε να επανέλθουμε για να ε, παρουσιάσουμε έκθεση πρόοδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την συζήτηση την οποία κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, μια δήλωση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση αντικτύπου ο Αντιπρόεδρος